στην ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων ε, Συγγνώμη, Κοινωνικών Ελευθεριών ε, και Δικαιοσύνης έτσι ώστε με τη σειρά της να μπορέσει στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας να το μελετήσει. Εμείς προτιθέμεθα να ψηφίσουμε